Perché... Συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. Παρακαλούσα και τους κυρίως δημοσιογράφους και φωτογράφους ε, να απελευθερώσουν εδώ το χώρο γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ε, σήμερα πρόκειται για μια μέρα πάρα πολύ σημαντική και δεν μπορούμε να δαπανούμε χρόνο. Αν κάποιος δεν ήταν ακριβής, ε, θα ήθελα να χαιρετήσω και να καλωσορίσω την ε, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την εκπρόσωπο της Ένωσης, γιατί παρουσιάστηκε εδώ στις 3 ακριβώς. Είναι η τρίτη φορά που η κυρία Άστον παρουσιάζεται εδώ ενώπιον αυτή τη Επιτροπή ε, και σήμερα με την παρουσία τη επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδουμε όλοι εμείς στο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό η σχέση αυτή να βασίζεται σε μια τακτική επικοινωνία γιατί όπως έχουμε πει ελοπίσαμε την ακρόαση της ε, Αντιπροέδρου και το Κοινοβούλιο θα διαδραματίζει το ρόλο του με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Και φυσικά ευχόμαστε σήμερα να υπάρξει μια σαφής αρχιτεκτονική της υπηρεσίας αυτής. Επίσης θα αξιολογήσουμε αν η πρόταση αυτή που θα παρουσιαστεί από την Αντιπρόεδρο θα λάβει να βάνει υπόψη τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και την εξουσία δημοκρατικού ελέγχου που του προσδίδεται από τη συνθήκη. Επίσης, στη συνεδρίαση αυτή έχουν ε, κληθεί και όχι μόνο τα μέλη της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά και από τις Επιτροπές Προϋπολογισμού Νομικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης Διεθνούς Εμπορίου, και Κομμάτων των Γυναικών και τα λέω αυτά για να μην πρέπει να ζητώ συγγνώμη κάθε φορά, αλλά θα πρέπει ε, αυστηρός ε, να διατηρήσω τον κατάλογο για όσοι ζητούν το λόγο και θα πρέπει να σεβόμαστε το χρόνο. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά αν δεν σέβεστε το χρόνο θα πρέπει να σας διακόπτω ενώ αναπτύσσετε τη, σχέση, τη σκέψη σας και την ερώτησή σας. και στο τέλος ε, της συνάντησης θα αφιερώσουμε 20-25 λεπτά στην ε, αποτιμήση της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών που έλαβε χώρα χθε. Αυτά είναι τα δύο θέματα που θα δούμε λοιπόν. Νομίζω ότι Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τις εργασίες σας και χωρίς χρονοτριβή να δώσω το λόγο στην ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κυρία Άστον. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι πάλι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα για να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και όπως σας είπα και ο πρόεδρος, θα σας ενημερώσω και για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που έγινε χτες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα μας που συζητήθηκε σε κοινή συνεδρίαση μεταξύ του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Υποθέσεων. Και πριν από δύο εβδομάδες στην Ολομέλη είχαμε τη Γενική Συζήτηση περί Εξωτερικών Υποθέσεων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε για την ενισχυμένη υποστήριξη που είχε η έκθεσή σας για την ΚΕΠΑ. Η δημιουργία υπηρεσία εξωτερικής δράσης παρουσιάζει μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη να οικοδομήσει κάτι το οποίο επιτέλους θα συγκεράσει όλα τα μέσα με τα οποία δραστηριοποιούμεθα. Όλα τα οικονομικά και επιχειρησιακά μέσα και μέτρα υπό μια κοινή στρατηγική. Τα... Οι λέξεις κλειδιά θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση των ευκαιριών και της ευελιξίας και όχι η επιβάρυνση με διοικητικά και γραφειοκρατικά μέτρα. Πιστεύω ότι η λογική που θα πρέπει να μας διέπει δείχνει ότι θα πρέπει η Ευρώπη να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο εξαιρετικά περίπλοκο όπου αλλάζει η ισορροπία των δυνάμεων. Η... Πάρα πολλά κράτη σήμερα είναι ευάλωτα. Κινδυνεύουμε από καταστροφές περιβαλλοντικές, από την παράνομη μετανάστευση. Οι κίνδυνοι επικρέμονται καθημερινά πάνω στη ζωή μας. Και γι' αυτό για να μπορέσουμε να συγκεράσουμε όλες, όλα αυτά τα θέματα και τους κινδύνους υπό ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο δημιουργούμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα προωθεί της, ε, τη γενική στρατηγική και τις επιμέρους πολιτικές. Συνδέοντας λοιπόν και συντονίζοντας τους διάφορους τομείς της πολιτικής θα αυξήσουμε το ευρωπαϊκό κύρος εάν εργαστούμε μέσα σε στεγανά, απομονώνοντας ε, τις πολιτικές μας κάτω υπό διαφορετική στρατηγική πτυχή, τότε δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και να ακουστεί η φωνή μας ε, τόσο δυνατά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προβάλλουμε εντονότερα την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, να είμαστε φιλόδοξοι και να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν και όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Σε Τότο σώμα πιστεύω ότι πάρα πολλά μέλη έχουν την ίδια προσέγγιση. Εκτίμησε ιδιαίτερα τη συζήτηση που είχαμε στην Ολομέλεια και το όραμα το οποίο προβλήθηκε για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πρέπει η Ευρώπη να δείξει την πυγμή τη στην παγκόσμια σκηνή και να ανταποκριθεί στις ευθύνες της για τη διεθνή και ευρωπαϊκή ασφάλεια. Καλύπτουμε ένα φάσμα εξωτερικών σχέσεων και δεν θα πρέπει τα διά, οι διάφορες διευθύνσεις και υπηρεσίες να αλληλοεπικαλύπτονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε το σημαντικό αυτό θέμα. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την διάσκεψη των Προέδρων όπου και το θέμα αυτό εφήγει θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω τις σαφείς μου απόψεις για την υπηρεσία αυτή και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχετε ενεργό συμβολή και συνδρομή για τη σωστή λειτουργία όχι μόνο στο θέμα του προϋπολογισμού αλλά και στο διοικητικό σκέλος, στο προσωπικό, στα στελέχη. Θα έχει λοιπόν το Κοινοβούλιο έναν εποπτικό ρόλο στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Οπωσδήποτε η υπηρεσία αυτή θα είναι υπόλογη όσον αφορά τον προϋπολογισμό της. Τον προϋπολογισμό της. Οι εξωτερικές δράσεις θα υπόκεινται στην ίδια μορφή δημοσιονομικού ελέγχου ως να ή το υπηρεσία της Κομισιόν. Τα στελέχη είτε προέρχονται από εθνικές ε, υπηρεσίες εξωτερικών, υπουργοί εξωτερικών, είτε προέρχονται από ευρωπαϊκά στελέχη, θα υπόκεινται σε έλεγχο ικανοτήτων και προσόντων και θα είναι υπόλογα βεβαίως στα πρότυπα του δημοσιονομικού κανονισμού. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε το, το αρνητικό επιχείρημα ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι λιγότερο ενωσιακή και ευρωπαϊκή από ό,τι άλλες υπηρεσίες. Θα βασιστεί στις ε, συνθήκες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και θα σέβεται απολύτως η υπηρεσία αυτή το κοινοτικό εκτιμένο και τις ευρωπαϊκές μεθόδους δεν είναι γενική διεύθυνση της Κομισιόν. Είναι όμως ε, διέπεται από τους κανονισμούς των γενικών διευθύνσεων της Κομισιόν. Όπως σας είπα, στα θέματα του προϋπολογισμού η επιρροή του Κοινοβουλίου θα αυξηθεί. Δεν υπάρχει πια συμφωνία κυριών που θα περιορίζει την επιρροή και την εποπτεία του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επικεφαλή των αντιπροσωπιών θα είναι στη διάθεσή σας για να αναφέρουν τα θέματα τα οποία αφορούν τις ε, χώρες τους και κάθε ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία θα έχει ένα στέλεχος επαφής, έναν αξιωματούχο επαφής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, οι επίσημες επισκέψεις θα ε, υποστηρίζονται από στελέχη από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ύπατοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να επισκέπτονται αυτήν την Επιτροπή και να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και το πρόγραμμά τους πριν διοριστούν επισήμως. Ε, συνάντησα τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στην Καμπούλ πρόσφατα, τον κύριο Βάιντα Σουσάκας, ε, σε θέματα Αφγανιστάν και μαζί με όλες τις ενέργειες πολιτικού ελέγχου θα συμβουλεύουμε τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα διαβουλεύουμε λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις βασικές πτυχές ε, της ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ξέρω ότι η αναπτυξιακή πολιτική θεωρείται σημαντική από πολλά μέλη του σώματος. Έχω προτείνει συγκεκριμένα προγράμματα δράσης για την υπηρεσία ώστε να ανταποκριθεί ακριβώς ε, στο έργο της εκεί που χρειάζεται, δηλαδή στην καρδιά της ευρωπαϊκής δράσης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος κατά την άποψή μου γιατί οι σχέσεις με ορισμένες χώρες πρέπει να είναι διαφορετικές από τις σχέσεις με άλλες χώρες. Αυτό το οριζόντιο γραφείο, η οριζόντια δρέωση αν θέλετε, η οριζόντια οργάνωση αποκρίνεται και στο πρότυπο της Κομισιόν. Ε, θα μπορέσει έτσι λοιπόν να έχει μια στρατηγική εποπτεία των διαφόρων ε, έργων και δράσεων. Πρέπει να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας σε πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο για να μπορέσει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Γι' αυτό η Υπηρεσία Εξωτικής Δράσης θα είναι υπεύθυνη για το στρατηγικό προγραμματισμό και θα έχει τη γενική εποπτεία. Για το, το ετήσιο πρόγραμμα και το εκτελεστικό και εφαρμοστικό πρόγραμμα είναι στα χέρια της Κομισιόν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα υπάρχει μετα, αντιμετώπιση ευθυνών. Εγώ θα βασίζομαι στον Άντρε Πίμπαλς για την ε, εξέλιξη και διαμόρφωση της πολιτικής καλής γυτνίασης. Και θα ακούω τη γνώμη όταν θα προετοιμάσουμε το στρατηγικό μας πρόγραμμα. Τέλος, οι προγραμματικές προτάσεις θα υποβάλλονται κοινώς θα προτείνω εγώ βεβαίως με τους αρμόδιους επιτρόπους στο σώμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα είμαστε ε, ε, από κοινού υπόλογοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι εσείς θα ασκείτε εποπτεία πάνω στο πρόγραμμα συνεργασία μας για την επιβεβαίωση της νομιμότητας της πολιτικής μας και αυτό το στοιχείο θα διατηρηθεί. Αφού αναφέρθηκα στη σημασία του ρόλου του Κοινοβουλίου, φυσικά να υπογραμμίσω ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι ο μόνος ε, εταίρος. Όπως είναι γνωστό, η δημιουργία της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ε, θα χαίρει τη υποστήριξη τη Κομισιόν και θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία στο Συμβουλίο των κρατών μελών. Το να εξεύρουμε συμφωνία μεταξύ των διάφορων πρωταγωνιστών δεν θα είναι κάτι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτό αν δείξουμε καλή θέληση και ευελιξία. Θα προτείνω στην Προεδρία όταν ε, κάθε θεσμός, κάθε όργανο θα έχει εξετάσει την νομική του πρόταση να συσταθεί το απαραίτητο πλαίσιο για διαπραγματεύσεις μεταξύ των τεσσάρων εταίρων, το Συνοβούλιο, το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και μου και όλα τα στοιχεία κλειδιά θα τεθούν επιτάπητο σε εκείνη τη συζήτηση. Συνάδελφοι, θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να καταλήξουμε σε ταχεία ολοκλήρωση, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα στα κρεμή ζητήματα. Σε, όλη αυτή τη σε όλα αυτά χρειάζεται συλλογική και συνεχή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, την Κομισιόν και με ανοιχτό διάλογο μαζί σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να το θέσω μα λέγεται υπηρεσία για ένα λόγο γιατί δεν θα βρίσκεται μόνο για να με επικουρεί αλλά για να βοηθάει και κυρίως την οικογένεια Ρέλεξ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού, Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συγγνώμη, φυσικά τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει για τα προγράμματα εξωτερική βοηθεία, για το σχέδιο οργανογράμματο, για ε, το προπολογισμό και για τι δομέ διαχείριση. Ευχαρίστω να απαντήσω στι ερωτήσει σα σήμερα και επίση να προωθήσω και τι προτάσει σα. Και θα ήθελα να κλείσω ευχαριστώντας τον κύριο Μπροκ και τον κύριο Φερχόφστατ για το χρόνο που μου έδωσαν στο να δούμε κάποιες από τις λεπτομέρειες για κάποια από τα θέματα που τους ανησυχούν ιδιαίτερα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Ήπατα πρόσωπο, η οποία και έφτασε εγκαίρως και σεβάστηκε και το χρόνο παρέμβασης. Ο γύρο ε, γύρος ε, συζήτησης προβλέπει να παρέμβουν οι συγητές των διάφορων επιτροπών. Καταρχήν ο κύριο Μπροκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να εφαρμόσει τη συνθήκη και να δημιουργήσει μια εξωτερική υπηρεσία ευρεία, η οποία να επιτρέπει ε, να μιλάει η Ευρώπη με μία φωνή. Η δυσκολία είναι ότι έχουμε δύο νομικές βάσεις, ε, την ε, κοινοτική και έχουμε και το Συμβούλιο, η συναπόφαση θα πρέπει να πραγματοποιείται όχι μόνο μεταξύ δύο θεσμικών οργάνων, αλλά μεταξύ τριών, το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Αναφέρατε μια σειρά θεμάτων για τον προϋπολογισμό, την απαλλαγή κλπ. Μήπως μπορείτε να είσαστε πιο ακριβείς στο θέμα αυτό. τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Κομισιόν θέτει ερωτήσει σχετικά με τον προπολογισμό και όσον αφορά τα δικαιώματα πολιτικού ελέγχου σε περιπτώσει ε, διοργανική ε, συμφωνίας ε, ή επιστολών. Σε πόσες λεπτομέρειες μπορούμε να μπούμε για να αποφύγουμε τα προβλήματα. Εάν πετύχουμε ομοφωνία στο θέμα αυτό, θα έχουμε όσον αφορά την υπηρεσία που όπως είπαμε θα πρέπει να είναι ευρεία, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος της κοινοτικής μεθόδου. Και γι' αυτό πολλές θέσεις της Κομισιόν ε, βρίσκουν κατανόηση σε εμάς. Θα θέλαμε όμως ε, να σας βοηθήσουμε να πετύχετε ε, και γι' αυτό ε, τίθεται το θέμα της εκπροσώπησής σας. Ποιος σας εκπροσωπεί όταν λείπετε, γιατί δεν μπορείτε να είστε πανταχού παρούσα. Πρόκειται οι επίτροποι θα ασχολούνται με τα κοινοτικά θέματα και από την πλευρά του Συμβουλίου ποιος θα σας εκπροσωπεί. Δεν θέλουμε να το κάνει αυτό ένας γενικός ε, διευθυντής, γενικός γραμματέας ή κάποιος άλλος υπάλληλος. Θέλουμε αυτό να γίνεται σε πολιτικό επίπεδο. Και τι γίνεται με το κυλιόμενο σύστημα των Προεδριών. Ευχαριστώ τον κύριο Μπροκ. Κύριος Φερχόφστατ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι για τη δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικής βάση πρέπει να τονίσουμε τρεις βασικές πτυχές. Πρώτον, ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η νομική βάση. Η πολιτικά και δημοσιονομικά, η απαλλαγή θα δίνεται από το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν αυτό να καλύπτεται από νομική βάση και ούτω να οριστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλε διευκρινήσει κλπ. Είναι σαφές. Απαλλαγή από εμά, από το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, η, η καλύτερη λύση είναι η υπηρεσία αυτή να είναι φιλόδοξη και να καλύπτει και πολιτικές όπως ανθρωπιστική βοήθεια, ανάπτυξη, πολιτική καλής γυτνίαση. Γιατί δεν είναι καλό να καλύπτουμε ας πούμε ανθρωπιστική βοήθεια με την εξωτερική δράση και όχι την πολιτική καλής γειτονίας. Ή θα έχουμε μια μικρή περιορισμένη υπηρεσία ανεξάρτητη από την Κομισιόν εξαιρετικά γραφειοκρατική με λίγο πολύ την οργάνωση του Ξαβιέ Σολάνα ή θα δημιουργήσουμε μια ευρεία ε, ε, μεγάλη εξωτερική υπηρεσία συνδεδεμένη με την Κομισιόν γιατί πρέπει να συνδεθεί με ένα θεσμικό όργανο που θα καλύπτει αυτές τις τρεις πτυχές. Και εγώ νομίζω ότι το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει μια ενισχυμένη, διευρυμένη εξωτερική υπηρεσία. Τώρα, Όσον, όσον αφορά ε, τους, αναπληρωτές, οι αναπληρωτές χρειάζονται διότι ε, είναι υπόλογοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ευχαριστώ τον κύριο Φερχώστα. Κύριος Ράκαμ για δύο λεπτά. Ραπκάι, συγγνώμη, για δύο λεπτά. Ja, hier sitze ich, wenn Sie mich suchen. Hier sitze ich, wenn Sie mich suchen sollten. Εδώ είμαι, αν ψάχνετε. Έχω κάποιες αμφιβολίες, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, πώς θα πρέπει να ξεκινήσω. Διότι όσον αφορά το δικό μου θέμα, το καθεστώς ε, του προσωπικού, δεν είναι κάτι το οποίο θα, βρει, θα συναντήσει γενική ικανοποίηση. Στην κυρία Αντιπρόεδρο είπα ότι θέλουμε να λύσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, θέλουμε να όσο γίνεται πιο γρήγορα τις εκκρεμότητες. Εάν επικαλούμαστε το πνεύμα της συλλογικότητα και διατυπώσουμε το ερώτημα, εγώ ξέρω αυτά που, είχαμε, που, που που εγκρίναμε στην έκθεση Μπροκ ε, πέρσι τον Οκτώβριο. Κανένας από την υπηρεσία σας ε, δεν ε, συνομίλησε μαζί μου, δεν ε, ήρθε σε επαφή μαζί μου για να ρωτήσει που μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να πει κανεί ότι η πρόταση δεν υπάρχει καν ακόμα. Όταν υποβληθεί επίσημα η πρόταση για τον κανονισμό του προσωπικού, τότε μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά υπάρχουν διάφορα πράγματα που έρχονται από διάφορες πηγές, κάποια έγγραφα, αλλά δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες. Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε λεπτομέρειες. Παρακαλώ όμως σύντομα να ξεκινήσει η συζήτηση για το που εσείς οι συνεργάτες, οι συνεργάτες σας, οι Κομισιόν, θα ασχοληθούν με αυτά που αποφασίσαμε πέρσι τον Οκτώβριο. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται, πότε μπορούμε να περιμένουμε την ε, τυπική πρόταση διότι όλους μας ενδιαφέρει να δημιουργηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ώστε να μπορεί να εργάζεται προς όφελες της κοινότητας. Θα πρέπει όμως να έχουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Ο κύριο Γκρέσλερ είναι στην αίθουσα, δεν τον βλέπω από εδώ και έχει ζητήσει το λόγο, εκπροσωπεί την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Όχι. Εφόσον λοιπόν απουσιάζει, Ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη, από προσωπεί την Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την υπατή ε, εκπρόσωπο. Όπως μπορείτε να δείτε από την έναρξη της συζήτηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι ισχυρό συμμαχός σας, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει σε μια ισχυρή υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης και δεν ε, σημαίνει ότι είναι ισχυρή αυτή η υπηρεσία θα σημαίνει κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για να διευρύνουμε για να αναπτύξουμε την κοινωτική μέθοδο. Πιστεύω παρόλα αυτά προκειμένου να μπορούμε να εξηγήσουμε την έννοια αυτή ενώπιον αποκλίνουσων απόψεων ε, μεταξύ κρατών μελών αφενός και κομισιών αφιταερού. Νομίζω ότι θα ήταν ε, καλό να έχει υπάρχει από πλευρά σας μια πραγματική διαθεσιμότητα για να αναλοποιηθεί ένα πολιτικό σύμφωνο με το Κοινοβούλιο. Ένα τέτοιο πολιτικό σύμφωνο σύμφωνα με κάποιες κατευθύνσεις γραμμές ε, που ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι συγητές ε, και αφορά τη νομική βάση και τον τρόπο με τον οποίο η σύνδεση με την Επιτροπή της ε, Αυτόνομης Δράσης θα λειτουργεί και αυτό αφορά και θέματα προπολογισμού και αφορά και αυτή τη διαπαφή που θα υπάρχει με την αναπτυξιακή πολιτική και αφορά και το θέμα και των αναπληρωτών. Συγκεκριμένα για τον προπολογισμό, εγώ μπορώ να πω ότι τα όσα είπατε είναι πολύ σημαντικά. Μπορεί να είναι και πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε το σημερινό προπολογισμό της ε, ΚΕΠΑ. Έχουμε μία δομή του προπολογισμού της ΚΕΠΑ που επιτρέπει να υπάρχει πραγματικός έλεγχος των μεμονωμένων αποστολών. Ευχαριστώ τον κύριο Κολτιέρη. Η κυρία Άστον για πέντε λεπτά τώρα έχει το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Μπροκ έθιξε το θέμα του ελέγχου του προϋπολογισμού που νομίζω ότι διευκρίνησε και ο κύριος Βερχόστατ χρησιμοποίησε τρεις λέξεις. Υπόλογος, ε, ε, προϋπολογισμός και απαλλαγή. Σύμφωνο και με τα τρία, με όλα αυτά. Όσον αφορά του πού είναι υπόλογη αυτή η υπηρεσία δημοσιονομικά, είναι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να το πω πιο, με πιο σαφή λόγια, πιο ξεκάθαρα. Δεν έχουμε απολύτως καμία διαφορά ως προς αυτό το αίτημα. Συμφωνώ κύριε Μπροκ με το ότι η Κομισιόν θα πρέπει να διατηρήσει τις ευθύνες ε, και τις αρμοδιότητές της. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου θεματοφύλακα αυτών των ευθυνών και οι ευθύνες είναι πάρα πολύ σαφείς. Το ερώτημα με τη δημιουργία αυτής της νέας υπηρεσίας είναι πώς να ξεκινήσεις όταν συγκεράζεις διάφορα στοιχεία εκπροσώπησης της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οργανώσεις, οι μη κυβερνητικοί οργανωσμοί, όλοι οι άλλοι φορείς το βλέπουν αυτήν την υπηρεσία ως μία ενιαία, μία υπηρεσία, ένα φορέα δηλαδή και πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά για να μην βλέπει κανείς τις ραφές αν θέλετε μέσα σε αυτό το ενιαίο μανδύα. Είναι λοιπόν ε, πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε σωστά. Όπως έχω δηλώσει και πολλές φορές στα μέσα ενημέρωσης, δεν μπορώ να είμαι ταυτόχρονα παρούσα σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σωστό σύστημα ε, εκπροσώπησης και αναπληρωτών αυτό πραγματικά είναι ένα κρεμέ ακο- ακόμα και θα το μελετήσω, θα σας ενημερώσω εγκαίρως και με συνέπεια πώς θα λειτουργήσει το σύστημα των αναπληρωτών, πώς, ποιος θα με αναπληρώνει. Δεν μπορώ δυστυχώς να είμαι τόσο πολλές φορές μαζί σας όσο θα ήθελα. Πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε ένα σύστημα αναπλήρωσης Θέλω να υπάρχει μία σωστή πολιτική εκπροσώπηση. Δεν θα πρέπει εμείς να αποτελούμε μία ε, μία ανταπόκριση στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από την συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα που είμαστε μέσα στο πλαίσιο της ε, συνθήκης, πιστεύω ότι η συνεργασία μας είναι εξαιρετικά ε, σημαντική και σημείωσα το μήνυμά σας ε, για την, το πολιτικό σας μήνυμα. Συμφωνώ με τον κύριο Βερχόφστατ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος σύστασης της υπηρεσία αυτής αν δεν είμαστε φιλόδοξοι στους στόχους μας. Θέλουμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα προβλήματα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ευημερία για τους πολίτες μας και ασφάλεια πρέπει αυτό να συμβαδίζει με την ευημερία και την ασφάλεια σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να απαγιώσουμε τις αξίες, τις πολύτιμες αξίες στις οποίες πιστεύουμε. Η πολιτική της καλής γυτνίασης βεβαίως θα αποτελεί μία από τις ε, πτυχές ε, της ε, υπηρεσίας αυτής. Πρέπει να βρούμε πώς θα το λύσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να έχουμε μία δύναμη δράσης έτοιμη να αντιδράσει στα προβλήματα εκεί και όπου παρουσιάζονται, όπου και όποτε παρουσιάζονται αυτό που πάρα πολύ με πιέζουν να κάνω είναι να προσδώσω μια γενική ευελιξία στη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας για να μπορέσουμε να παρεμβαίνουμε γρήγορα. Θα μιλήσω μαζί σας βεβαίως και με τα θέματα της τελέχωσης, με την ίση μεταχείριση, με την ε, ελάχιστη απλούστευση ε, των διαδικασιών. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, πώς θα επιλέγονται τα στελέχη και όλα τα συνεφή. Κύριε Γκαλτιέρη, μιλήσατε για ε, ένα πολιτικό σύμφωνο. Βεβαίως, είναι σαφές ότι η πολιτική είναι η κατευθυντήρια γραμμή και θα έχετε οπωσδήποτε το δικαίωμα εξάστηση των πολιτικών σας αρμοδιοτήτων επί της υπηρεσίας αυτής. Ευχαριστώ την κυρία Αντιπρόεδρο. Εσείς ε, πραγματικά σέβεστε το χρόνο που έχει χορηγηθεί στον καθένα. Ελπίζω να το σεβαστούν και οι βουλευτές. Ο κύριος Σαλαφράνκα, ευχαριστώ. Στην πρώτη σας ε, εμφάνιση βάση ε, δεσμευτήκατε ότι η ΚΕΠΑ θα είναι ένα βιβλίο που θα το γράψουμε από κοινού και εσείς δώσατε την εντύπωση που δώσατε. Σήμερα το πρωί με κάποιους φίλους, εγώ σχολίασα αυτό που είχε πει ο Όσκαρ Βάιλτ, θα το πω στα αγγλικά, ποτέ δεν έχει κανείς ε, μια δεύτερη ευκαιρία για μια πρώτη εντύπωση για να δημιουργήσει πρώτη εντύπωση. Πέρα από το ότι είναι πολύ ευφύ η φράση αυτή, κυρία Άστον, θέλω να σα πω ότι όμω ε, η εντύπωση μπορεί να αλλάξει και μπορεί να βελτιωθεί. Και εγώ νομίζω ότι μια χρυσή ευκαιρία για να γίνει αυτό είναι ακριβώ αυτό το θεμελιώδε κεφάλαιο του βιβλίου, όπω είπατε εσεί σήμερα το απόγευμα, η δημιουργία δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Εσεί ε, σήμερα το απόγευμα αναλάβατε σημαντικέ δεσμεύσει ε, πολιτική, πολιτική και μολυτικό και δημοσιονομικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δώσατε και ένα καλό μήνυμα ε, λέγοντας ε, ότι να παρουσιαστούν ε, ή επικεφαλής ε, ε, των ε, της Ουάσιγκτον και της ε, Καμπούλ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως, να σκεφτούμε και το εξής. Εμείς δεν θέλουμε να δοθεί ουσιαστικά μία μάχη για την εξουσία από τα κράτη-μέλη στα πλαίσια αυτής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Θα θέλαμε εμείς να υπερασπιζόμαστε εδώ το κοινοτικό συμφέρον και θα ήθελα να μου απαντήσετε στο θέμα των ε, μεταφορών ε, ενέργεια, μετανάστευση, τι συγκεκριμένε διευκρινήσει για το χρονοδιάγραμμα, πότε θα παρουσιάσετε τι προτάσει σα και αν ο Γενικό Γραμματέα και δύο ε, αναπληρωτέ γενικοί γραμματεί, όπω ρώτησε ο κύριο Φερχόφστατ, ε, θα είναι πολιτικέ προσωπικότητε. Ευχαριστώ. E κύριος ένα μισή λεπτό δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θα περάσω απευθείας στην ερώτηση. Κυρία Άστον, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν ενθαρρυντική, θα έλεγα. Υπάρχουν ακόμα κάποιες λεπτομέρειε που θα πρέπει να συζητήσουμε, έχω ερώτηση όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού. Καθότι αυτό είναι ευαίσθητο θέμα, όχι μόνο για τα κράτη-μέλη, αλλά και για εμά ω εκπροσώπους ε, των ε, Ευρωπαίων πολιτών, πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε την σωστή γεωγραφική εκπροσώπηση στο προσωπικό της νέας υπηρεσία Η δίκαιη κατανομή των θέσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα για τα νέα κράτη-μέλη και τα μικρά κράτη-μέλη. Αυτό είναι κάτι απόλυτα μετρήσιμο αφού θα έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη του προσωπικού. Πώς μπορείτε λοιπόν να διασφαλίσετε την δίκαιη κατανομή των θέσεων, όχι μόνο όσον αφορά τον αριθμό, αλλά και το επίπεδο εκπροσώπησης. Ε, είναι μιλάμε για εκπροσώπηση των κρατών μελών, αλλά και των διπλωματών των κρατών μελών. Και επίσης, ε, τον ειδικό απεσταλμένο ε, Συμπεριλαμβάνεται αυτό στο οργανόγραμμα. Ε, πρόσφατα επισκεφτήκατε έξι υπουργού εξωτερικών. Έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε υπουργού εξωτερικών ω ειδικού απεσταλμένου, γιατί εμεί δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι καλή ιδέα. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατακαιρματισμό τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Το λόγο έχει Λάστοφ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχετε μία... Έναν απίθανο ρόλο. Πρέπει να κάνετε και εξωτερική πολιτική και να ε, φτιάξετε αυτή την υπηρεσία. Πραγματικά δεν σας ζηλεύω να τα κάνετε όλα αυτά δε ταχύτατα. Σας ευχαριστώ που αναφέρατε τις ε, προτεραιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς αυτή την υπηρεσία. Έχω δύο-τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, πώς εξασφαλίσετε τη συνοχή και προς τον συνάδελφο Σαλαφράνκ ήθελα να πω ότι δεν χρειαζόμαστε ένα παντοδύναμο γενικό γραμματέα αλλά μια δυνατή ομάδα από ανθρώπους η οποία θα, επιβάλλει τη θα... θα εξασφαλίσει τη συνοχή. Δεύτερον, τα σημεία συνάντησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες ε, της Κομισιόν. Η κομβική σύνδεση δηλαδή με την Κομισιόν. Είπατε ότι με τον αρμόδιο επίτροπο θα φέρετε το θέμα στο κολέγιο των επιτρόπων. Εσείς θα αποφασίσετε εν τέλει ποιος έχει τον τελευταίο λόγο. Ή ε, το κολέγιο των επιτρόπων, εσείς ή, ή, ή από κοινού, μαζί και τα δύο σκέλη. Τρίτη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι ένας συνδυασμός ε, και προς τα έξω, αλλά και ε, εν μέρη Υπουργείο Άμυνας. Έχει θέματα Υπουργείου Αμήνης και εξωτερικής πολιτικής. Θα ήθελα λοιπόν να μου διευκρινίσετε πώς θα μοιράσετε αυτές τις αρμοδιότητες μεταξύ άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Ευχαριστώ, η συνάδελφος Μπραντνερ, για ένα μισή λεπτό. Um, you know, I could this... Ευχαριστώ. Με, με, κάλυψε ο συνάδελφός μου, κύριος Λάμστορφ, στα περισσότερα που ήθελα να πω και γι' αυτό θα ήθελα να σχολιάσω ένα κείμενο το οποίο επισήμως δεν το έχουμε. Η κορεπέρ, ε, από την Κορεπέρ το έχω αυτό το οργανόγραμμα. Αλλά επισήμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν το έχει. Θα ήθελα λοιπόν ε, δεδομένου ότι μέχρι τώρα έχουμε το Συμβούλιο όσον αφορά τις, ε, τις αποστολές στο Κωσυφοπαίδιο, εν συνεχεία στην Κομισιόν έχουμε τις διάφορες αποστολές ε, στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Ωραία, μπορούν να συντονιστούν όλα αυτά, αλλά κάτω από ένα κοινό πλαίσιο δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την δομή του Συμβουλίου και εν συνεχεία μέσω του Γενικού Γραμματέα να του δώσουμε άλλο ένα παντοδύναμο μέσον, ένα όργανο στα χέρια του, την εξωτερική υπηρεσία, ε, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Με τις ε, νέες εξελίξεις και τις νέες δομές στη γραμματεία του Συμβουλίου τα πράγματα δεν έχουν διευκολυνθεί καθόλου, το αντίθετο. Λοιπόν, αντί δεν θέλω επίσης από την πλευρά της Κομισιόν να έχουν ένα μπλοκ επιταγών και να γράφουν επιταγές και δεν είναι λεφτά. Θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε μια σωστή δομή η οποία θα συγκεράσει αυτά τα δύο σκέλη. Θα ήθελα λοιπόν τα, τις παρατηρήσεις σας. Επίσης, εάν για κάθε αποστολή θα υπάρχει μία γραμμή στον προ, προϋπολογισμό. Αποστολή Β, Γ, Δ. Ευχαριστώ κύριε Στάνο για ένα μισή λεπτό. Μικρόφωνο παρακολουθούμε. Εμείς... Θα στηρίξουμε τις ε, προκλήσεις σας ε, όσον αφορά τη δημιουργία του, της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Είμαστε όμως και ρεαλιστές και γι' αυτό στηρίζουμε το σημείο 14 του πρωτοκόλου της Λισαβόνας που λέει ότι δεν θα δοθούν νέε αρμοδιότητες όσον αφορά την ΚΕΠΑ ή την ΕΠΑ μετά την Λισαβόνα. Πιστεύουμε ότι οι εξωτερικές υποθέσεις και τα θέματα άμυνας θα πρέπει να παραμείνουν κυβερνητικά με ομοφωνία και θα πρέπει να ηγηθείτε εσείς ε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ε, το Κοινοβούλιο ε, έχει περισσότερες αρμοδιότητες τώρα και έχει αρμοδιότητες όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τον κανονισμό του προσωπικού. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο επικροτεί τη δυνατότητα ελέγχου και του δημοκρατικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και επίσης έχουμε το δικαίωμα συνένεση σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες επικροτούμε την ε, σύμφωνη γνώμη της ε, Επιτροπής μας της ε, ΑΦΕΤ όσον αφορά τους εκπροσώπους. Έχουμε όμως κάποιες ανησυχίες όσον αφορά το μοντέλο Brock η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία αυτή δηλαδή να εμπίπτει στην Κομισιόν παρά να είναι ξεχωριστή η υπηρεσία με δικό της προϋπολογισμό. Γι' αυτό σας ρωτάμε ποιο είναι το πρότυπο που προτιμάτε εσείς και πιστεύετε ότι και τι πιστεύετε θα γίνει με την πρόταση του κυρίου Μπροκ όσον αφορά την ΚΕΠΑ και την ΕΠΑ. Ευχαριστώ τον κύριο Πάνο και Μέγερ για λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Άστον Ξέρετε, αρχικά η κοινοβουλευτική μου ομάδα ήταν ε, ιδιαίτερα επικριτική με την αρχιτεκτονική αυτή τη υπηρεσία εξωτερική δράση, γιατί περιλαμβάνει την, αρχιτεκτονική την ασφάλεια, την ανάπτυξη, τη συνεργασία, την πολιτική γειτονία και από τη δική μα σκοπιά θα έπρεπε να ε, αποκλείεται το, να αποκλείεται από αυτό το όραμα της ασφάλειας. Όμως τα πράγματα έχουν ως έχουν πέρα από τη δική μας θέση. Εμείς θα θέλουμε τελικά να θέσουμε τέλος ε, σε αυτό το προσωρινό χαρακτήρα γιατί αφενός έχουμε ε, πρόβλημα με το καταστατικό τη στιγμή της πρόληψης των εργαζομένων γιατί δεν ξέρουμε αν είναι καθορισμένο ή όχι. Έχουμε πρόβλημα οργανογράμματος και αρμοδιοτήτων και εγώ νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να απαντηθεί το συντομότερο. Όταν, όσο αυτό δεν το προσεγγίζουμε εντάχει, νομίζω ότι αντί να μιλάμε, όπως και σήμερα, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για την επίσκεψή σας στην Μέση Ανατολή, που είναι πράγμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα προβληματισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους επίκους στην Ιερουσαλήμ και τα λοιπά, ε, εξακολουθούμε να μιλάμε για θέματα που αφορούν προβλήματα στις αρμοδιότητες. Και εγώ νομίζω ότι ε, θα έπρεπε και σύμφωνα με τη γνώμη της δική μας ομάδας να αντιμετωπίσουμε ε, άμεσα όλα αυτά τα ζητήματα. Επίσης, στήθηκε το θέμα του ελέγχου της υπηρεσίας. Όπως ξέρετε, στον 20ο αιώνα ε, δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη για να ελέγχουν τα εθνικά κοινοβούλια την πολιτική ασφάλειας και διακόπτει ο πρόεδρος τον ομιλητή. Δυστυχώς ε, δεν ε, ολοκληρώσατε μέσα στο χρόνο που σας είχε δοθεί η αντιπρόεδρος. Όχι, δεν είναι ακόμα η σειρά σας. Ο κύριος Μπαλίτερ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και σας κύριε Αντιπρόεδρε. Το ουσιαστικό θέμα είναι εάν παρουσιάζεται παρουσιάζεστε εξ ονόματος του Συμβουλίου ή εξ ονόματος της Κομισιόν. Διπλό καπέλο. Στο τέλος ένα καπέλο θα έχετε και το άλλο θα κρέμετε στην καρδερόμπα. Λοιπόν, ε, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή το ρεύμα σας πρόχνει προς την Κομισιόν. Εσείς τι θα προτιμούσατε, πού θα προτιμούσα θα προτιμούσατε να ήσασταν, κάπου στη μέση θα είναι η χειρότερη λύση. Τι γίνεται με την ισορροπία δυνάμεων. Ένα θεσμικό όργανο, δύο θεσμικά όργανα. Το προσωπικό, τα στελέχη που θα υπηρετήσουν σε αυτήν την υπηρεσία δεν θα πρέπει να φοράν δύο καπέλα, πρέπει να ξέρουν που ανήκουν. Και ο λόγος τώρα στην Αντιπρόεδρο, 7 λεπτά. Δύσκολο να τα καταφέρετε, αλλά αν είστε τόσο καλοί όπως και πριν θα τα καταφέρετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω. Μάλιστα κύριε Σαλαφράγκα, δεύτερη ευκαιρία για να κάνει κανεί μια πρώτη καλή εντύπωση, υπομονώ και για την τρίτη, Καθώ ε, θα γράφω αυτό και το κεφαλαίο του βιβλίου. Δεν νομίζω ότι βλέπω εδώ να υπάρχει ε, ένα, μια άνηση μάχη των κρατών μελών ε, και εγώ χαίρομαι που εκπροσωπώ τα συμφέροντα τη κοινότητα γιατί προέρχομαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά τι πολιτικέ ενέργεια μετανάστευση και μεταφορών η Κομισιόν Λοιπόν, με, την, με τις αρμοδιότητές της επιβλέπει όλες αυτές τις πολιτικές και φυσικά θα υποβάλει αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είχα μία πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή πρόσφατα από τον κύριο Καλές για το πώς ε, θα εργαστούμε ε, από κοινού για το θέμα, για οποιοδήποτε είδο θέμα, είτε μιλάμε για τις τα κτλ. Και η υπηρεσία απάντησε σε αυτόν εξ ονόματος του Επιτρόπου. Όμως τελικά υπάρχει γενικό συντονισμό. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο και βέβαια θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία τώρα οι γραμματείς και οι γενικοί αναπληρωτές, εμείς θεωρούμε ότι ε, οι άνθρωποι αυτοί θα αποτελούν ε, ουσιαστικά ε, την υπηρεσία, μάλλον τους ανθρώπους που στελεχώνουν την υπηρεσία της εξωτερική δράση. Τώρα αναφερθήκατε επίση στη γεωγραφική κάλυψη. Εγώ προσπαθώ συνεχώ να παρακολουθώ κάνουμε, κατέστησα σαφέ ότι θα πρέπει να έχουμε μια υπηρεσία που να εκπροσωπεί την Ευρώπη. Έτσι, λοιπόν, όλα τα κράτη-μέλη, όλοι θα πρέπει να αισθάνονται ότι ε, υπάρχει ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ε, όμω χρειάζεται χρόνο για να το πετύχουμε αυτό. Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει επιθυμία να εκπροσωπούμαστε καλύτερα στι υπηρεσίε που θα δημιουργήσουμε και θα το πετύχω αυτό, όμω θα χρειαστεί κάποιο χρόνο πρέπει να το παρακολουθούμε και επίσης θέλω να διασφαλίσω ότι θα έρχονται άνθρωποι όχι μόνο επικεφαλής των αντιπροσωπιών, αλλά και μεσαία στελέχη προκειμένου να κερδίσουν την κατάλληλη εμπειρία, να αποκτήσουν την κατάλληλη εμπειρία για να γίνουν επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Όμως θα το φροντίσουμε. Τώρα, για του υπουργού εξωτερικών και του ειδικού απεσταλμένου, δεν είχα αυτό κατά νου. Ε, έχω μια συνάντηση με όλου του ειδικού απεσταλμένου αυτή την εβδομάδα, νομίζω, για να μου πούν τι ακριβώ ε, κάνουν και θα επανέλθω σε εσά. Ε, είχαμε περισσότερο αυτό το θέμα με, το, με τα ταξίδια. Αν παραδείγματο χάρη κάπου δεν βρίσκομαι εγώ, αλλά βρίσκεται ο υπουργό εξωτερικών, μπορεί να με εκπροσωπήσει. Κυρία Λάμστορφ, είναι αδύνατη δουλειά αυτή, αλλά εδώ είμαι ακόμα και την κάνω. Ε, τώρα η μία φωνή είναι να λένε όλοι το ίδιο πράγμα, σαν να είναι η δική μου φωνή. Συμφωνώ ότι ε, πρέπει να ε, με κρίνουν, όμως θα πρέπει και να υπάρχει και κατάλληλη διαχείριση και δίκηση της υπηρεσίας από τον αρμόδιο. Το Σώμα των Επιτρόπων θα λάβει τις τελικές αποφάσεις ε, για θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες κομισιών. Όπως κάνει συνήθως, οι προτάσεις θα γίνονται από κοινού, αλλά το Σώμα των Επιτρόπων θα λαμβάνει τις αποφάσεις, τίποτα δεν αλλάζει. Επίσης, σε αυτή την, εξωτερική, σε αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ε, ελπίζω θα μπορέσουμε να τροφοδοτούμε και με θέματα που συμβαίνουν εκεί επί τόπου, θα διατηρούμε φυσικά ενημερωμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι και πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιε είναι οι αρμοδιότητες του καθενό Τώρα, η πρόληψη ε, των σειράξεων, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εκεί που διαφωνούμε είναι ότι εγώ δεν θέλω να συστήσω ένα τμήμα, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι θεμελιώδες θέμα ε, που πρέπει να αντιμετωπίσει η υπηρεσία, είναι οριζόντιο και όχι κάθετο ζήτημα νομίζω ότι πρέπει να, να το δούμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό σκέλος των όσων κάνουμε αλλά ε, καλύπτει και ένα μεγάλο τμήμα του έργου μα, Γιατί αν δείτε λόγω χάρη τι συμβαίνει στη Σομαλία, τι προσπαθούμε να κάνουμε και για την καταπολέμηση της παρετίας. Ε, το έργο μα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει και αναπτυξιακό έργο επιτόπου και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την μεταβατική κυβέρνηση, το κράτο που χρειάζεται περισσότερη βοήθεια, προκειμένου να μπορέσει να προσφέρει ασφαλεία στους πολίτε του. Όλα αυτά θα μπορούσα να πω ότι συνάδουν προς την πρόληψη της σύρεξης. Έχουμε την πρόληψη, το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά θα ε, εντάσσονται στο έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Τώρα για τον Γενικό Γραμματέα ποιος ξέρει ποιες εθνικότητες θα είναι. Τώρα κύριε Τάνεκ, ε, εγώ ανέφερα ότι υπάρχει ένα σύνδεσμο ε, με την Κομισιόν. Υπάρχει ούτω ή άλλω ένα αυτόματο σύνδεσμο. Αλλά αν δημιουργήσω την υπηρεσία στην οποία πιστεύω εγώ, η συνθήκη απαιτεί και νομίζω θέλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το εξή. Πρέπει να είμαστε επιτόπου προκειμένου να μπορέσουμε να δείχνουμε ότι είναι ενδράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάποια μέρη μπορεί να δίνεται έμφαση στο εμπόριο, αλλού στην κλιματική αλλαγή, αλλού να έχουμε άλλα θέματα όπως η Σομαλία να χρειάζονται ε, στρατιωτικές δράσεις. Αυτά θα τα δούμε και ορισμένα είναι αρμοδιότητες Κομισιόν. Έτσι λοιπόν ο σύνδεσμος με την Κομισιόν πρέπει να είναι σαφής. Το πώς το προσδιορίζουμε αυτό και το πώς το διαρθρώνουμε θα πρέπει να το σκεφτούμε. Αλλά εγώ είμαι σαφής. Δεν ε, θέλουμε να αφαιρέσουμε το ρόλο των ε, επιτρόπων αλλά και επιτόπου θα ε, υπάρχει ε, ανάληψη δράση και όσοι εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα θα καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Κύριε Μαϊέρ, σε ό,τι αφορά τώρα την πρόσληψη υπαλλήλων, νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε για το πώς ε, θα προχωρήσουμε στο μέλλον δεν έχει συσταθεί ακόμη και δεν λειτουργεί ακόμη η υπηρεσία. Ε, όμως ε, σεβόμαστε το χρονοδιάγραμμα ε, και να σας πω ότι δεν έχω μια υπηρεσία για να γράψει ε, όλα τα έγγραφα, να συντάξει όλα τα έγγραφα και να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Εγώ ελπίζω ότι τελικά ε, θα μπορέσουμε να συστήσουμε αυτή την υπηρεσία και θα μπορέσετε να υποστηρίξετε αυτό το έργο και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα σας ικανοποιήσει για τη Μέση Ανατολή. Θα αναφερθώ σε αυτό σύντομα, είναι πολύ σημαντικό. Και τέλος, ε, για το θέμα της επιλογής μεταξύ Κομισιού Συμβουλίου, ε, κοιτάξτε, πρέπει η Άγκυρα να είναι και στα δύο. Πρέπει να είμαστε σταθεροί και στα δύο. Ευχαριστώ την κυρία την Πρόεδρο. Κύριε Τάνοκ, θέλετε το λόγο. Διαδικαστικό δεν μου απαντήσετε για το αν οι εξωτερικές υποθέσεις θα έχουν την πρωτιά, θα, είναι δηλαδή επικεφαλής. Νομίζω ότι απάντησα νωρίτερα. Η ΚΕΠΑ είναι σαφής, όπου τα κράτη-μέλη έχουν τις ευθύνες τους και είχαμε κάνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς θα μοιράσουμε τους Κύριε Τάνοκ, ε, σας έδωσα το λόγο, αλλά δεν μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε αυτό κάθε φορά. Το λέω για τους υπολείπους. Ε, ε εντάξει, να το λάβετε υπόψη. Αυτό δεν μπορείτε να ξαναπέρετε το λόγο συνεχώς. Τώρα, μετά την παρέμβαση των συζητών έχουμε τους εκπροσώπους ε, που, των επιτροπών που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα συζητούσα να μην κάνετε εισαγωγέ και να κάνετε μία και μόνο ερώτηση. Ζολή, ένα λεπτό. Κύριε την Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Ανάπτυξης, της οποίας προεδρεύω, θα ήθελε μια και μονο ερωτηση ζωλη ενα λεπτο κυριε προεδρε κυριε προεδρε η επιτροπη αναπτυξη τη οποια προεδρευω θα ηθελε μια απαντηση στην εξής απαντήσει, η συνθήκη τη Λισαβόνα προσδιορίζει την αναπτυξιακή συνεργασία ω αυτόνομη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη οποία ο κύριο στόχο είναι η μείωση και η εξάλληψη τη φτώχεια. Ε, έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε ποιε είναι οι ανάγκε των πληθυσμών και όχι ποια είναι τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ βλέπετε το ρόλο τη αναπτυξιακή πολιτική στο πλαίσιο τη εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ μπορείτε να εγγυηθείτε ε, ότι δεν ε, θα ε, καλύπτει άλλες ζητήματα πέρα από την εξάλληψη της στόχιας. Ε, η δική μου η Επιτροπή θα ήθελε να σας καλέσει για μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Θα έχετε μια τέτοια πρόσκληση. Ευχαριστώ την κυρία Ζουλή. Τζαραντήλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ απλή ερώτηση για την κυρία Άστον για το ποιος ε, ε, ε είναι υπεύθυνο γιατί. Θα μπορούσατε να μας επιβεβαιώσετε ότι η εξωτερική υπηρεσία θα σεβαστεί τις αρμοδιότητες ε, του Επιτρόπου αρμόδιου για εμπορικές υποθέσεις όπως, ορίζεται, ε, όπως λειτουργεί δηλαδή η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και το, όπως ορίζει το άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Δηλαδή, πιστεύετε ότι το εμπόριο και, και τα, οι εμπορικές διευθύνσεις θα πρέπει να ανήκουν στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κάλφιν για ένα λεπτό. Κυρία, είπατε αρμοστή, εδώ είμαι, ναι. Είπαμε ότι δεν θα, υπάρχει, δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των εφορετικών υπηρεσιών. Σωστό. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να γίνουν μεταφορές ε, στον προϋπολογισμό από την Κομισιόν στην υπηρεσία και από το Συμβούλιο στην υπηρεσία. Επίσης, όσον αφορά την απαλλαγή και την ευθύνη, είπατε ότι η, η γενική ιδέα είναι να ε, διαιρέσουμε το γενικό πρόγραμμα με τις εξωτερικές υποθέσεις από τη μία πλευρά και την υλοποίηση στην Κομισιόν από την άλλη πλευρά. Ποιος, οπότε, ποιος θα είναι υπεύθυνο ε, ε, οικονομικά, οικονομικά, δημοσιονομικά, ποιος θα είναι υπεύθυνο η υπηρεσία της Κομισιόν ή η δική σας υπηρεσία και εσείς ίδια. Και, οπ, διακόπτει ο Πρόεδρος. Μπράνερ για ένα λεπτό. Μη σας κάνει εντύπωση κι εγώ έχω δύο καπέλα. Ε, ε έντομες ερωτήσεις. Ε, συμφωνείτε με την ποσόστοση του ενός τρίτου στις ε, υψηλές θέσεις και Μήπως είσαστε υπέρ, πέρα από το, το mainstreaming για την ισότητα των δύο φύλων, ε, πιστεύετε να υπάρχει και συντονισμός στα υψηλά επίπεδα, διότι εγώ δεν πιστεύω στο mainstreaming εάν δεν υπάρχει και κάποιος υπεύθυνο γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπράντνερ. Αυτό είναι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Αντιπρόεδρε, ε, έχουμε συζητήσει για το θέμα του mainstreaming ε, σε επιτροπή ε, στην πράξη τι μορφή θα έχει αυτό. Τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πράξη, στις εξωτερικές σχέσεις, πώς θα εφαρμοστούν δομικά. Ε, τι δομή δηλαδή θα έχουμε για το mainstreaming των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποτελούν ε, σημαντικό κομμάτι όλων των εξωτερικών σχέσεων και όλων των αποστολών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Άντελο. κύριος Ντανζέν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω για την πτυχή της διαχείρισης των κρίσεων και της απάντησης της κρίσης, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της αξιοπιστίας της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Έχετε στη διάθεσή σας στρατιωτικά μέσα που μπορούν να ενεργοποιηθούν για να ε, δοθούν απαντήσεις και αντιδράσεις ε, στις φυσικές καταστροφές, όπως είχαμε στην ΑΕΤ, όμως αυτό θα πρέπει να γίνει ε, ουσιαστικά χωρίς να υπάρχει γραφειοκρατία ε, και θα ήθελα να τοποθετηθείτε σε αυτό και επίσης θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα μέσα ε, της ε, Κομισιόν για την απάντηση στις κρίσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Ντανζέν. Σε αυτό το σημείο θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Άστον για να απαντήσει, αν είναι δυνατό, σε πέντε λεπτά. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Ζολή, για την ανάπτυξη, για την εξάλληψη της στόχιας. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι ένας κοινό στόχος. Η διαφορά που ελπίζω να επιφέρουμε είναι ότι θα βρούμε καλύτερα μέσα και θα βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιφέρουμε αυτή την κατάσταση, αυτή την πρόοδο δηλαδή της καταπολέμησης και εξάλληψης της φτώχειας. Όταν ήμουν υπεύθυνη ε, επίτροπος για το εξωτερικό εμπόριο και βλέποντας την κατάσταση στην ΑΕΤ σήμερα, πιστεύω ότι παρουσιάζεται μια θαυμάσια ευκαιρία να συγκεράσουμε τις ενέργειές μας για την επίτευξη του τελικού στόχου. Δηλαδή θα δώσουμε μια νέα όθηση και θα υπάρχουν και καλύτερα μέσα επίτευξης. Όσον αφορά το εμπόριο, η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου πιστεύω ότι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου <laughs> σας τα έχει πει αυτά, σας έχει βάλει να ρωτήσετε, να θέσετε αυτές τις ερωτήσεις. Και η απάντησή μου είναι ε, σαφώς, ε, ναι, βέβαια, βέβαια. Όμως θα πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα αυτά που γίνονται επί του εδάφους. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμός. Όμως θα είναι ε, δική μου ευθύνη να το συζητήσω αυτό με τον αρμόδιο επίτροπο. Αυτός είναι υπεύθυνο, ο Καρλ Ντεγκούχτ. Ως τον κύριο Κάλφιν για το προϋπολογισμό. Ως αντιπρόεδρος είναι σαφέστατο ότι έχω ευθύνες, είμαι και επίτροπος βεβαίως. Είναι η Κομισιόν για τον προγραμματισμό που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον προγραμματισμό. Η Κομισιόν δεν αλλάζει τίποτα. Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τα θέματα του δημοσιονομικού ελέγχου, απλώς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργούν ακόμα πιο αποτελεσματικά στο μέλλον. Και η κυρία Μπράτνερ, μόνο ένα τρίτο δεν αρέσουν το, το 1 τέταρτο, το 1 τρίτο, δεν μου αρέσουν τα τέταρτα μερίδια. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, για όλα τα κράτη-μέλη, αφορά όλα τα κράτη-μέλη, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανισορροπίας της διάστασης του φύλου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπερισχύει το αντρικό φύλο σε όλες τις υπηρεσίες οριζοντίες και καθέτος και γι' αυτό πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Βεβαίως, σε όλα τα κράτη-μέλη το έχω πει αυτό και στις διπλωματικές υπηρεσίες. Θέλω να κάνω κάτι θετικό για τη διάσταση του φύλου και για να επιβληθεί μια καλύτερη ισορροπία. Η κυρία Χότλερ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα. Βεβαίως, θα αποτελέσουν μέρος και του προγράμματος κατάρτισης, έτσι ώστε όλοι να καταλάβουν ότι αποτελεί και αυτό μία οριζόντια διάσταση. Ε, συνειδητοποιώ ότι έχουμε το διάλογο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεχίζεται με ορισμένε χώρε. Ε, δεν ξέρω αν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο θα ήθελα να είναι. Εγώ θέλω να αποτελέσει βεβαίω βασική πολιτική και διάσταση που να υπάρχει παντού. Και είμαι δεσμευμένη προς αυτό το στόχο. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, διαλέγοντας καλύτερα τα θέματα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε στις σχέσεις μας ή να αποσαφηνίσουμε ορισμένα θέματα τα οποία είναι συγκεχημένα. Ιδίω με την Αμερικανική πλευρά και με την Χίλαρη Κλίντον νομίζω ότι πολλά περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. κύριος ένα από τα θέματα που μου είπαν σαφώς από στατιωτικής πλευράς είναι να η αλυσίδα ανάθεσης εντολών να είναι σύντομη. Η, κάθετη δηλαδή απο, οργάνωση των λήψης αποφάσεων να είναι σύντομη. Όταν ήμουν στην ΑΕΤ είδα ορισμένα θαυμάσια παραδείγματα ε, ε, της διοικητικής μέρημνας και πώς δίνονταν οι διάφορες εντολές και πώς ήταν οργανωμένη από στρατιωτικής πλευράς η διοικητική μέρημνα έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις συναφείς υπηρεσίες, ε, την πυροσβεστική, τις νοσοκομιακές υπηρεσίες κλπ που χρειαζόντουσαν για να επιτελέσουν το έργο τους, το, το ανθρωπιστικό. Δηλαδή η διοργάνωση της ε, γραμμής ε, εντολών ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική και όλη η ανάθεση της διοικητικής μέρημνας. Πολύ ωραία. Ας έρθουμε τώρα στο κύριο της συζήτησης που αφορά τους σκιώδεις, Θα ξεκινήσει ο κύριος Βόμποντα με ένα λεπτό στη διάθεσή του. Ευχαριστώ. κύριο Γκουαλτιέρη πήρε το λόγο και μου ζήτησε να επανέλθω στο ε, βασικό ερώτημα της Επιτροπής αυτής. Αναφερθήκατε στο, στους γενικούς ε, διευθυντές και αναπληρωμένες και γενικούς διευθυντές ε, των διαφόρων υπηρεσιών. Ε, εντάξει, ε, είπατε ότι ε, θα εμπιστευτείτε τους υπουργούς εξωτερικών να κάνουν κάποιες δηλώσεις στο όνομά σας. Α, καλή τύχη στο να τους ελέγξετε. Αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου, συμπεριλαμβανομένου εντός του Κοινοβουλίου όπου θα ζητάμε πολιτική εκπροσώπηση στο όνομά σας, υπό τον έλεγχό σας, σε, διάλογο με εμά. Αυτό πρέπει να το σκεφτείτε πολύ προσεκτικά. Και ε, τελευταίο θέμα, ε, κυρία Άστον, ελπίζω να συμφωνήσετε ότι για τους πολίτες εντός της Ευρώπης και για τους πολίτες εκτός της Ευρώπης θα πρέπει να αναγνωρίσουν ε, ότι υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική. Το αν αυτή προέρχεται από το Κοινοβούλιο ή από, την, ε, ή το Συμβούλιο, αυτό δεν είναι σημαντικό. Για μας είναι, για, για τους έξω δεν είναι. Αλλά εσείς θα πρέπει να διασφαλίσετε να υπάρχει μία φωνή όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική για την, κοινωνική, για την κοινή αναπτυξιακή πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σπόποτα, κυρία Νέιτς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, κυρία ε, είπατε εκπρόσωπε. Ε, εδώ βρίσκομαι, καλό απόγευμα. κοιτώ τα τελευταία έγγραφα, άσχετα από την πηγή τους, είτε προέρχονται από την ε, Κομισιόν, από το Συμβούλιο, από τι υπηρεσίε από το Κοινοβούλιο, μπορώ μόνο να ε, συμπεράνω ότι ε, πολλή πρόοδος έχει σημειωθεί και έχουμε τουλάχιστον πιο σαφή εικόνα των πραγματικά δύσκολων θεμάτων τα οποία πρέπει ακόμα να λυθούν. Ένα από αυτά είναι η σχέση ανάμεσα στις ε, πολιτικές ε, στρατιωτικές ε, δομές και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Καταλαβαίνω ότι ο στρατιωτικός τομέας ή πρώην στρατιωτικός τομέας θέλει να διατηρήσει μικρές σύντομες αλυσίδες εντολών, αλλά εσείς θα είσαστε τελικά υπεύθυνοι. Πώς το προβλέπετε αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν μπορείτε να το αφήσετε αυτό να ξεφύγει από τα χέρια σας εμείς να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Λούνατσεκ, ένα λεπτό. Κυρία Άστον, θα ήθελα να επανέλθω στα θέματα που ήδη έθιξαν ο κύριος Λάμστορ και η κυρία Μπραντνερ σχετικά με την ΚΕΠΑ που αποτελεί μέρος ενός οργανογράμματος το οποίο, το οποίο επίσημα δεν έχουμε. Ε, εδώ γίνεται αναφορά όχι όμως ως ε, κομμάτι του συνολικού συστήματος και πολλοί από εμά πιστεύουμε ότι αυτό είναι λάθος τρόπος να γίνει αυτό. Η ε, συνθήκη της Λισαβόνας έχει την αντιμετώπιση των κρίσεων και τα θέματα αυτά σαν μέρος του συστήματος. δεν θα πρέπει να ξεχωρίσει το κομμάτι. Μερικοί από εμά εδώ πέρα θα, αντιτεθούμε στην, στον προπολογισμό της Κομισιόν ε, διότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι. Μπορείτε να μας απαντήσετε αν θέλετε να το διατηρήσετε έτσι ή αν θέλετε να ακολουθήσετε την επιθυμία του Κοινοβουλίου, να αποτελούν αυτά ένα απόσπαστο κομμάτι της ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σπορέμπε για ένα λεπτό, πρόεδρε, εκπρόσωπο. Υπάρχει ισχυρό κίνδυνο ότι τα νέα κράτη-μέλη θα υποεκπροσωπούνται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και ήδη το βλέπουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εντυπωθεί περισσότερο ε, στα πλαίσια της ε, περαιτέρω ε, διαδικασίας πρόσληψης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στις άλλες διπλωματικές υπηρεσίες. Υπάρχουν 130 ε, αντιπροσωπείες σε όλο τον κόσμο. Πόσοι επικεφαλείς ε, αντιπροσωπείων θα προέλθουν από τα νέα κράτη-μέλη προβλέπετε. Είπατε επίσης ότι θέλετε γεωγραφική κάλυψη ε, στο θέμα της πρόσληψης και θα το πετύχετε. Αλλά πώς θα το πετύχετε και πώς σχεδιάζετε να το πετύχετε και πώς ε, θα εξεύρετε την ισορροπία που επιθυμούμε εμείς στα κράτη-μέλη να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική δράση; Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πορέμπα. Σούλτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Άστον, συμφωνούμε γενικά οι πολιτικές ομάδες ότι η εξωτερική η υπηρεσία θα υπόκειται στον πλήρη έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πανέρχομαι στο βασικό ερώτημα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα αναλάβετε εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και μεμονωμένων κρατών μελών. Παραδείγματο χάρη, ε, πυρηνικός αφοπλισμός, πολιτική της Μέσης Ανατολής και ούτω καθεξής. Πού βλέπετε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εάν υπάρχει διάσταση απόψεων. Πώς θα προβάλλετε αυτή την κοινή ευρωπαϊκή θέση, την κοινή ευρωπαϊκή γνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόλτς. Ο κύριος Προβέρος, πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόσωπε. εγώ θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι η αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί ε, σωματωμένο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής, ε, συναφές τμήμα και επομένως η συνάφεια μεταξύ αυτών των δύο πολιτικών θεωρείται κάτι θεμελιώδες. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, εσείς ε, θεωρείτε ότι η υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης ε, που θα θέτει σε εφαρμογή την εξωτερική πολιτική θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες και στην αναπτυξιακή πολιτική και αν έπιασε αρμοδιότητες. Τελευταία ερώτηση. Μέσω ποιων εργαλείων εσείς σκοπεύετε να συνεργαστείτε με τον αρμόδιο για την ανάπτυξη επίτροπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Προβέρα. Το λόγο τώρα έχει αντιπρόεδρος Άστον για πέντε λεπτά. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σβόμποντα, αναφερθήκατε στο ρόλο του Γενικού Γραμματέα και των, εξωτε... Υπουργών Εξωτερικών, αν μπορώ να τους ελέγξω. Very, very helpful in two ways. One... αλλάζοντας λοιπόν καπέλο, πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ ε, ε, συνεργάζονται πάρα πολύ καλά και χρήσιμοι ε, οι γενικοί γραμματείς όταν έχουμε πάει μαζί σε αποστολή ε, το έχουν, κάνει, έχουν διαβιβάσει τα μηνύματά μας πάρα πολύ καλά και πολλές φορές αναγκάστηκαν να με αντικαταστήσουν να κάνουν μια ομιλία όταν εγώ δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα Βεβαίω, ε, σημείωσα τι παρατηρήσει από χτέ για την πολιτική εκπροσώπηση ε, και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και μέσω Συμβουλίου και Κομισιόν αλλά το Συμβούλιο δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική εκπροσώπηση θα βρούμε έναν τρόπο όπως είπαμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η πολιτική ασφάλειας και η εξωτερική πολιτική να ε, ε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μέσω της υπηρεσίας εξωτερικών, ε, εξωτερικής δράσης. Το θέμα κλειδί είναι ο συντονισμός που πρέπει να επιτύχουμε. Πολλοί, πολλά μέλη ρώτησαν πώς θα επιτευχθεί αυτός ο συντονισμός. Βεβαίως, ανάλογα με τις συνθήκες, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία κρίση, όταν πρέπει να διαχειριστούμε μία κρίση τα πράγματα στην ΑΕΤ, ήταν διαφορετικά και διαφορετικά πρέπει να αντιδράσουμε, ε, ενώ στη Χιλή πάλι ήταν μία άλλη κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες και το θέμα είναι ακριβώς να συντονίσουμε και να επιλέξουμε τις καλύτερες ενέργειες. Γι' αυτό οι δράσεις μας πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αλλά και να ταιριάζουν, να είναι κατάλληλες για τις συγκεκριμένε συνθήκες. Η κυρία Λίβτσεκ για τη διαχείριση κρίσεων. Βεβαίως αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών μας. Ένα διάγραμμα είναι διάγραμμα και Έστω και τρισδιάστατο πάλι είναι διάγραμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι θα πρέπει να είναι κανείς σε θέση να το περιγράψει πολύ συγκεκριμένα. Με όποιον τρόπο και αν προσπαθήσεις να το ενσωματώσεις σε μία δομή πρέπει να ανταποκρίνεται στην, σε μία ανταπόκριση την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε, να παρουσιάσουμε. Παραδείγματο χάρη στην ΑΕΤ, στη Βοσνία, η αντίδρασή μας είναι διαφορετική. Άρα λοιπόν το διάγραμμα αυτό δεν θα είναι διαφορετικό, ο τρόπος αντίδρασης θα είναι διαφορετικός. Ο τρόπος ανταπόκρισης καλύτερα. Τώρα, δεν θα σας δώσω συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για τη στελέχωση της υπηρεσίας, ε, ανάλογα με το κάθε κράτος μέλος. Εγώ απευθύνθηκα σε, σε όλα τα κράτη-μέλη για να μου πούν τη γνώμη, της, τη γνώμη τους. Σας είπα ότι εγώ θέλω τα καλύτερα στελέχη, θέλω να περάσει η διάσταση του φίλου, να υπάρχει μια ισορροπία βεβαίως και θα αρχίσουμε την επιλογή το, του προσωπικού. Όμως χρειαζόμαστε και ορισμένο χρόνο γιατί δεν μπορούμε αμέσως στον πρώτο γύρο να τα κάνουμε άλλα. Όλα. Συγκεκριμένου αριθμού, πόσου θα πάρουμε από πού. Όμω ε, γνωρίζω το θέμα και ήδη έχω λάβει πάρα πολλά, ε, πάρα πολλά βιογραφικά για προσλήψεις. Τώρα πώς θα συγκεράσουμε τις επόψεις εκεί όπου υπάρχουν διαφορετικές ε, γνώμες. Τώρα αφορά το καπέλο του Συμβουλίου. Καταρχάς πρέπει στα πλαίσια του Συμβουλίου να καταλήξουμε σε αποφάσεις και σε συμπεράσματα. Αυτό είναι σαφές. Π.χ. η πολιτική της Μέσης Ανατολής. Εδώ έχουμε μια ισχυρή εξωτερική πολιτική και μπορώ να δράσω πιο αποτελεσματικά. Βεβαίως θα υπάρχει διάλογος, βεβαίως θα υπάρχει συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Όμως πρέπει να εμπλουτίσουμε την, ε, το πλαίσιο της ε, ΚΕΠΑ δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλο τον κόσμο. Και η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να συνεργάζεται με την εξωτερική πολιτική. Αυτό που θέλω να εξασφαλίσω είναι ότι γίνεται στην εξωτερική πολιτική να ταιριάζει βεβαίως να ανταποκρίνεται αντίστοιχα σε πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Στο σημείο αυτό έχουμε προβλέψει τις ε, παρεμβάσεις ε, Κοιτάξτε, έχουν ζητήσει 25 άτομα το λόγο, πρέπει να δημιώσω στο μισό τον αριθμό αυτό. Φυσικά θα λάβω υπόψη το που ανήκει ο καθένας και τη σειρά με την οποία ζήτησε ο καθένας το λόγο. Αν η κυρία Αντιπρόεδρο συμφωνεί στο σημείο αυτό, για να επιτρέψουμε να γίνει διάλογος με τους συναδέλφους, δεν θα έλεγα να συζητήσουμε το δεύτερο θέμα που έχουμε προβλέψει στη Μερσία Δάταξη, δηλαδή την σύνοψη της έκβασης της συνεδρίας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο κύριος Μάουρο, τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Στον, θα ήθελα την άποψή σας για την θεσμική ισορροπία που ε, θα αφορά τις αποφάσεις της υπηρεσίας που σας προεδρεύετε. Δηλαδή να εξηγήσω, ως είπατε εκπρόσωπος εσείς μαζί με τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής πρέπει να τύχετε ψήφου έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της προσωπικής ακρέωσης. Δεν σας φαίνεται τώρα το ως ε, ανομαλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να έχει μόνο μία συμβουλευτική εξουσία όταν μιλάμε για τη σύσταση νομοθεσίας για μία υπηρεσία η οποία θα εξαρτάται από εσά άμεσα και δεν αναφέρομαι στο θέμα του προπολογισμού και του καταστατικού αλλά στο τμήμα της οργάνωσης και της λειτουργίας της υπηρεσίας. Ευχαριστώ τον κύριο Μάουρο. Ο κύριο Κόπα για ένα λεπτό. Κύριε Κόπα μάλλον. want to my voice. Θα ήθελα κι εγώ να ενώσω τη φωνή μου με όλες τις επιφυλάξεις που ακούσατε μέχρι τώρα για τη γεωγραφική ε, εκπροσώπηση. Προερχόμενο από μια μικρό, μικρή χώρα, την Ελλάδα, θα ήθελα σε αυτό το οργανόγραμμα να υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπερισχύσουν και πάλι οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα αντιμετωπίσετε, τις, ε, πώς εξασφαλίσετε μια δίκαιη κατάσταση μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών. Επίσης, Ποιους, ε, ε, ποια στελέχη θέλετε να υπηρετούν στην υπηρεσία από το δημόσιο, μόνο διπλωμάτες, άλλοι αξιωματούχοι. Ευχαριστούμε κύριο Σπρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μία και μόνο ερώτηση. Πότε πιστεύετε, κυρία Άστον, ότι θα ε, καταστεί επιχειρησιακή αυτή η υπηρεσία, δηλαδή από ποια ημερομηνία και πέρα θα μπορούμε να πούμε ορίστε υπάρχει υπηρεσία και δεν μιλάμε μόνο για κάτι που θα είναι επί χάρτου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε πιτα. που, που μιλήσατε και τόσο σύντομα. Ευχαριστώ. Λέω ο κύριο Δεν καταλαβαίνω. Δεδομένου ότι πρέπει να κάνουμε οικονομίες, πώς θα μπορέσετε να επιβάλλετε την δημοσιονομική ουδετερότητα. Εγώ θα σας υποστηρίξω, αν θέλετε αυτό, να το επιβάλλετε βεβαίως. Εμείς, ως αν αγόρια και άντρες βεβαίως καταλαβαίνετε ότι μας αρέσουν πάρα πολύ τα οργανογράμματα. Αλλά θέλω να ρωτήσω για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ε ψηλά στην προτεραιότητα θα είναι, χαμηλά στο οργανόγραμμα θα, θα είναι. Και πώς θα αντιμετωπίσετε και την ε, ΚΟΟΜ. Ευχαριστώ τον κύριο Χόιτ. Κόβαξ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Lady Άστον. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, έχετε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο μπροστά σας για την ε, δημιουργία αυτής της ε, ισχυρής υπηρεσίας. Είπατε ότι θέλετε να τη στελεχώσετε με διπλωματικό προσωπικό και βεβαίως θα πρέπει να επιτευχθεί στην εκπροσώπηση μια γεωγραφική ισορροπία. Χάρηκα που είπατε ότι είσαστε αποφασισμένοι να το κάνετε και να εδραιώσετε μια γεωγραφική υπηρεσία μεταξύ των κρατών μελών. Πιστεύω ότι αυτό το στοιχείο πρέπει να περιληφθεί στο καταστατικό του προσωπικού, η αρχή δηλαδή και της γεωγραφικής ισορροπίας αλλά και της διάστασης του φύλου να ε, υπάρχουν, να αναφέρονται στο καταστατικό. Όσον αφορά τις αποστολές σε τρίτες χώρες, εκεί όπου ήδη υπάρχουν υπηρεσίες δικές μας, θα μειώσετε το τοπικό προσωπικό ή θα αυξήσετε τους διπλωματικούς υπαλλήλους, τι θα κάνετε. Μάλιστα, ας δώσουμε το δικαίωμα απάντηση στην κυρία Την Πρόεδρο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μάουρα, ελπίζω να καταστεί σαφέ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει την ευθύνη για όλα τα θέματα του προπολογισμού, έτσι όπω το περιέγραψα. Συγγνώμη αν δεν ήμουν σαφή, αλλά την ε, χρηματοοικονομική ευθύνη για τα δημοσιονομικά θα την έχει το Κοινοβούλιο. Τελεία. Δηλαδή, Εμεί, θα πρέπει να έρθουμε εδώ να λογοδοτήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θα κάνουμε σε εσωτερικό επίπεδο. Κυρία Κοπά, για το θέμα τη κυριαρχία των μεγάλων κρατών. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια κυριαρχία των μεγάλων κρατών πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ουσιαστικά θα έχουμε εκπροσώπηση όπως έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή θα έχουμε ε, και ισορροπία σε ό,τι αφορά τα δύο φύλλα κτλ. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι είναι οι εθνικοί τους διπλωμάτες και, αυτοί, και αυτά θα υποβάλουν τα βιογραφικά και τελικά θα ακολουθηθεί μια διαδικασία για την πρόσληψη. Όμως τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν ποιον θέλουν να στείλουν. Εγώ ζητώ το καλύτερο, τους καλύτερους. Αυτό με ενδιαφέρει. Κύριε Πρέτα, για την ημερομηνία θα έχουμε μια σταδιακή διαδικασία. Έχουν τεθεί όλες οι προθεσμίες για το Συμβούλιο προκειμένου να ληφθούν οι αρχικές αποφάσεις εγκαίρων. Θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει το δικό του έργο και θα τεθεί σε λειτουργία η υπηρεσία, Όμω όλα αυτά θα γίνουν σταδιακά γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ε, θα προσλάβουμε και του κατάλληλου ανθρώπου για το μέλλον και φυσικά θα πρέπει να ε, παρακολουθούμε συνεχώ το θέμα για να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί καλά η υπηρεσία σε ό,τι αφορά την ιδιαιτερότητα του προπολογισμού. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ μαζί σα. Αν μείνουμε τώρα στην ιδιαιτερότητα του προπολογισμού θα έχουμε ε, δύο άτομα σε κάθε την προσωπία και τελικά εγώ δεν θα μπορέσω να κάνω όλα όσα θέλω να κάνω. Το ξέρουν αυτά τα κράτη-μέλη. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, όμω αν μα υποστηρίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό θα είναι ουσιώδε και θα σα εγγνωμονώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θέλω παντού να υπάρχει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ε, θέλω και περισσότερη υπερογνωμοσύνη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μου αρέσει να συζητώ για το πώς θα διασφαλίσουμε ε, ότι αυτό θα αποτελεί τιμήμα των δράσεων όλων. Ήμουν ε, υπουργό αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ξέρω πόσο σημαντικό είναι να μην ε, είναι ο μόνο άνθρωπο που θα ασχολείται με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όλοι θα πρέπει να ασχολούνται μέσω και τη κατάρτιση, μέσω του συστήματο. Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι καλύπτεται το θέμα αυτό και σκέφτομαι ήδη από τώρα πώ θα δράσουμε καλύτερα για να πετύχουμε αυτό που το οποίο συμφωνούμε να Αναφερθήκατε στην αρχή της γεωγραφικής ισορροπίας και στην ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις. Νομίζω ότι αυτό θα υπάρχει ούτως ή άλλως και να μειώσουμε τον αριθμό του τοπικού προσωπικού. Ε, το προσωπικό επιτόπου εκτιμάται ιδιαίτερα από τις ε, αντιπροσωπείες κομισιών γιατί έχει πολύ μεγάλη και τα κτλ. Δεν θέλω να δώσω το λάθος μήνυμα, θέλω ε, ουσιαστικά όμως να αντικατοπτρίζουμε αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει δηλαδή σε όλα τα ζητήματα που φύγουν τις χώρες τις οποίες θα έχουμε παρουσία Ευχαριστώ την κυρία Αντιπρόεδρο και να μπούμε στο δεύτερο γύρο. Ένα λεπτό παρακαλώ έχετε. <clears throat> Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για τα όσα είπατε όσον αφορά την γεωγραφική ισορροπία. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω ότι ναι, οι χώρες θα πρέπει να στείλουν τους καλύτερους υποψηφίους. Δεν έχει τεθεί εκ των προτέρων προφίλ. Ίσως όμως να πρέπει να έχει κανείς σε συγκεκριμένο προφίλ για να μπορεί να χειριστεί κρίσεις και Και θα ήθελα να αναφερθώ και στο άλλο θέμα που αναφέρατε. Θα ήθελα να ακούσω πώς βλέπετε την πρόταση να υπάρχουν τρεις αναπληρω... αναπληρωτές και πώς ε, συνδέεται αυτό με θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Ευχαριστώ. Άτκινς για ένα λεπτό. Πρόεδρε, πριν ξεκινήσω μπορεί να θίξω ένα διαδικαστικό. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ρωτήσουμε ε, σχετικά με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, μας τελειώνει ο χρόνος. Είχαμε σκεφτεί να μην ε, κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για να μην μπερδέψουμε τις, ε, τις δύο συζητήσεις. Δεν έχουμε χρόνο, έτσι λοιπόν θα σας ζητούσα να πάρετε το λόγο να αποθετείτε το πρώτο σημείο, το άλλο θα το δούμε σε άλλη συνεδρίαση. Κυρία Άστον, ε, υπάρχει η ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετράει πια σε σχέση με τη Ρωσία ή την Κίνα. Και το 2009 η ομάδα διεθνούς κρίσης είπε ότι η Ευρώπη θα δείξει το βάρος της μόνο με καλύτερο συντονισμό και εκμεταλλευόμενη ε, ε, ε, στο βαθμό που είναι δυνατόν τα μέσα που έχει στη διάθεσή της τη διπλωματία, την ε, αναπτυξιακή βοήθεια και, την, ε, το στρατό. Ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα το καταφέρει αυτό δεδομένη της δυσκολίας να συμφωνήσουν μεταξύ τους οι Υπουργοί της Ευρώπης σε, για οποιοδήποτε θέμα. Πόσο μάλλον που αντιμετωπίζουμε κάποιες, ε, κάποια πολύ δύσκολα θέματα όπου κανένας δεν φαίνεται να έχει διάθεση να αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Πώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Ε, ευχαριστώ. Βέμπερ, για ένα λεπτό. Λέει Άστον, ένα από τα θέματα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η παρακολούθηση εκλογών είναι μια χρονοβόρος και ακριβή διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σαφώς μεγάλη διαφάνεια όταν γίνονται τέτοιες ε, ενέργειες. Ε, όχι μόνο για τις συγκεκριμένες εκλογές, αλλά για όλη την ε, περιφέρεια. Θα ήθελα λοιπόν ποια προτεραιότητα θα δώσετε αυτά τα χρόνια στην παρακολούθηση εκλογών από ευρωπαϊκούς παρατηρητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Βέμπερ. Ο Γιάννης, ο οποίος είναι πρόεδρος της διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπιών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Στον, ε, μιλήσαμε για το τρίγωνο Κομισιόν Κοινοβούλιο Συμβούλιο. Μέσα στο Κοινοβούλιο φαίνεται να αναπτύσσεται μια αποτελεσματική διπλωματία. Υπάρχει και ο θεσμός της διάσκεψης των Προέδρων των ε, Αντιπροσωπιών και μπορώ να σας πω ουσιαστικά αποτελούν το ένοπλο σκέλος του εξωτερικού της εξωτερικής πολιτικής. Είναι ένα μέσο που ε, εσείς θα πρέπει να το έχετε κατά νου και για το μέλλον. Είμαστε 40 ε, άτομα και πάνω και εμείς ε, θα μπορούσαμε να έρθουμε σε συντονισμό και με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή αλλά και με εσά για να αναπτύξουμε αυτή την πολιτική. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τη συνεργασία με αυτό το θεσμό. Ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη. Σάιρους Βόσκη για ένα λεπτό. Uh, thank you, uh, Mrs. Ashton. Ευχαριστώ κύριε Άστον. Έχω μία ερώτηση. Πώς μία εκπρόσωπος θα είναι. Είπατε εκπρόσωπος όταν το γραφείο της δεν είναι εκπρόσωπος δεν εκπροσωπεί τους 27, τις 27 χώρες, μεγάλες, μικρές, μεσαίες. Την περασμένη φορά στο Στρασβούργο είπατε ότι θα επικρατήσει αξιοκρατία, σαν να μας εξασφαλίζει αυτόματα η αξιοκρατία και την θεμητή ισορροπία. η εκπροσώπηση, σωστή εκπροσώπηση βασίζεται στην νομιμότητα και στην αξιοπιστία. Η νομιμότητα οδηγεί στην ισχύ, στη δύναμη. Δεν θέλουμε να είμαστε δυνατοί. Άρα λοιπόν η γεωγραφική ισορροπία δεν θα πρέπει να είναι μία απλή υπόσχεση, αλλά θα πρέπει να είναι μία δεσμευτική πολιτική. Έχουμε γεωγραφική ισορροπία, πρέπει να υπάρχει γεωγραφική ισορροπία και στην ευρωπαϊκή διπλωματία, εφόσον υπάρχει αυτή η γεωγραφική ισορροπία και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν και στα άλλα θεσμικά όργανα. Συγγνώμη, δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουν όλοι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα δώσουμε για πέντε λεπτά το λόγο στην κυρία Στον για να απαντήσει. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επρίσια, ε, ε, συγχωρήστε με αν δεν πρόφερα σωστά το όνομα μάλλον δεν το πρόφερα σωστά, τα γεωγραφικά θέματα, όπως θα πω ε, ε, επανειλημμένα στην ε, συζήτηση αυτή, βρίσκονται πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξή μου. Καταλαβαίνω τα, τις ανησυχίες, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι να εκπροσωπήσετε σωστά. Θα πρέπει να περιμένετε να δείτε τα αποτελέσματα. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι είμαι απόλυτα σαφής για το θέμα αυτό και καταλαβαίνω ότι αν αναζητούμε έναν εμπειρογνώμονα σε συγκεκριμένο τομέα, δεν είναι τυχαία επιλογή. Όταν σας λέω στείλτε μας τους καλύτερους, ενώ για τη συγκεκριμένη δουλειά. Για παράδειγμα, ε, μπορεί οι ικανότητες, τα προσόντα που χρειάζονται να είναι διαφορετικά ε, για μια αποστολή στη Γεμένη από ότι για μια αποστολή ε, στην Κίνα. Τα δέχομαι όλα αυτά. Απλά είπα ότι πραγματικά θέλω τους καλύτερους. Διότι για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα θα χρειαστεί δημιουργικού ανθρώπου που είναι διατεθειμένοι να ανοίξουν νέου δρόμους. Αυτό θέλω. Όσον αφορά τους τρεις ε, αναπληρωτές. Έχει γίνει η πρόταση και έχουμε αρχίσει να τη συζητάμε. Άλλα θεσμικά όργανα θα έχουν σαφείς θέσεις. Εγώ απλά λέω ότι θα πρέπει να δημιουργήσω μηχανισμό το θέμα της ε, πολιτικής εκπροσώπησης ε, πολύ σωστά τέθηκε και το δέχομαι απόλυτα. Το πώς θα φανεί αυτό θα πρέπει να το διαπραγματευτούμε. Και όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, αυτό θα το εξετάσουμε μαζί με τον Επίτροπο Oettinger ε, υπό το του δικού του ρόλου και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Κύριε Άτκινς, αυτό που είπατε είναι σημαντικό το αν η συνοχή που προτείνουμε θα έχει σημαντικότερο αντίκτυπο στις στρατηγικές μας ε, σχέσεις με την ε, Ρωσία, την Κύρια και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ε, δυνατότητές μας να ενεργήσουμε επιτόπου. Εγώ θα έλεγα ναι και να σας, πάρω ένα πολύ, να δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα των όσων έχουμε ήδη δει. Η θέση των 27 κρατών μελών για τη Μέση Ανατολή στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου του 2008 έγιναν δεκτά και όπου και να πήγα στο Ισραήλ και στον αραβικό κόσμο ε, έγιναν ε, αποδεκτά και αυτό είναι πολύ καλό εργαλείο για μένα για να ενεργήσω επί τόπου. Πιστεύω ότι τα διάφορα στοιχεία της ε, υπηρεσίας μας θα σημάνει σημαντική διαφορά. Οι Παλαιστίνοι θα χρειαστούν δυνατότητα οικοδόμησης δυναμικού και είναι πολύ σημαντικός και εδώ η Ευρώπη έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Και νομίζω επίσης ότι η δυνατότητα να εκπροσωπούμε ε, την Ευρώπη ένα άτομο στο ε, κουαρτέτο είναι πολύ σημαντικό. Αναγνωρίστηκε η συμβολή μας ε, και αναγνωρίστηκε από το Ηνωμένα Έθνη, τις Ηνωμένε Πολιτείε και τη Ρωσία. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα του τι θέλω να κάνω όσον αφορά την παρακολούθηση των εκλογών. Ε, κυρία Βέμπερ, ναι, χρειαζόμαστε περισσότερη ορατότητα, δεν ξέρουμε ακόμα πώς να το κάνουμε αυτό, αλλά έχετε πολύ δίκιο ότι κάνουμε πολλή δουλειά, απομένουν πολλά να γίνουν όμως. Επικροτώ. Αυτούς που συμμετείχαν σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών ε, δέχομαι τις θέσεις ε, του πώς μπορεί να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικά στο μέλλον. Όσον αφορά τις διακοινοβουλευτικές ε, ε, σχέσεις, είναι πολύ σημαντικές διότι ε, συμβάλλει στην πρόθεση των διμερών μας σχέσεων. Ε, λέω λοιπόν ότι αν μπορώ να υποφεληθώ από τις εμπειρίες σας ε, θα το κάνω για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Κύριε Σαρισβόλσκι, γεωγραφική ισορροπία, δεν θέλετε να είναι μονολόγια. Ναι, σίγουρα. Ναι, με τους 27 επιτρόπους είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Στην υπηρεσία θέλω να βεβαιωθώ στο χρόνο να υπάρχει γεωγραφική ισορροπία. Ξέρω ότι υπάρχουν θέματα όπου πολλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι δεν υπάρχει επαρκή ισορροπία και θα τη διορθώσω αυτή. Δεν θα υποσχεθώ όμως συγκεκριμένε θέσεις σε συγκεκριμένες χώρες, ούτε θα υποσχεθώ να λύσω το πρόβλημα μιας μεμονωμένης χώρας με τη μία. Θα το κάνω όμως το χρόνο και σας υπόσχομαι θα το πετύχω. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, ας περάσουμε στο Catch the Eye, κύριο Σεβερίν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχετε διπλή εκπροσώπηση Κομισιόν και Συμβούλιο και τριπλή νομιμότητα Συμβούλιο, Κομισιόν και Κοινοβούλιο δεν πιστεύετε ότι αυτοί που υποτίθεται ότι πρέπει να σας εκπροσωπούν, δηλαδή πληρωτές αυτοί, θα πρέπει να έχουν ε, την ίδια πολλαπλή νομιμότητα και δυνατότητα εκπροσώπησης. Και αν το πει κάποιος ότι αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη, εγώ θα απαντούσα ότι ούτε απαγορεύεται όμως από τη συνθήκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σεβερίν. ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω για την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πολυμερή φόρουμ και στον ΟΗΕ ιδιαίτερα, ειδικά. Ε, πέρσι μάθαμε από την αντιπροσωπεία μας ότι η ο πρέσβης μας πρέπει να εργαστεί ενώ δεν είχε σαφείς εντολές από τις Βρυξέλλες. Έχουμε λοιπόν μεγάλες προκλήσεις ε, τώρα που εφαρμόζεται η συνθήκη δεδομένου ότι τα μέσα στη διάθεσή μας είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Επίσης, διάφορα όργανα εμπίπτουν σε διαφορετικές αρμοδιότητες Εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το καθεστώς του παρατηρητή θα, θα, θα ήθελα να ξέρω πώς θα αντιμετωπίσετε το πλέγμα αυτό των, των σχέσεων. Ευχαριστώ κύριε Αντρική. Είμαι ο κύριος ένα λεπτό. Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα. Όσον αφορά την προσπάθειά μας να ορίσουμε πολιτικούς αναπληρωτές, μήπως μπορούμε να εφαρμόσουμε το άρθρο 33 για να το επιτύχουμε. Δεύτερον, συγκρίνοντας τώρα την προσέγγιση του Συμβουλίου ως προς την εδραίωση της υπηρεσίας αυτής με την προσέγγιση της Κομισιόν, Ποια προσέγγιση πιστεύω ότι δημιουργεί τις περισσότερες ε, ανησυχίες. σας προβληματίζει περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Τάφ. Βαν για ένα λεπτό. Καλό σας απόγευμα, Βαρονάστον. Να χαίρομαι που ακούω τις τελευταίες δύο ώρες ότι όλα είναι σημαντικά, όμως το πρόβλημα είναι η φιλοδοξία για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τελικά να απορροφήσει τις εθνικές ε, πρεσβείες. Αυτό είναι ένας πραγματικός κινδύνος ε, καθώς ήδη τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν πολύ μεγάλους προϋπολογισμούς και αυξάνονται ακόμη και το Βρετανικό Foreign Office είναι υποχρηματοδοτούμενο αυτή τη στιγμή. Είπατε ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε την υπηρεσία ως μια γενική διευθύνση της Κομισιόν. Αυτό θα μας μας μας αν ο ρόλος της υπηρεσίας ήταν απλώς ε, παρήχε ανθρωπιστική βοήθεια και οικοδόμηση μετά τη